Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μια άλλη περίπτωση τώρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Καμπότζη, το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Που τη βλέπω, η κυρία Λοχμπίλερ δεν έχει έρθει. Και συντάκτης. Οπότε, δίνω τον λόγο στον κύριο Ουιασντόφσκι. Έχετε τον λόγο. pani przewodnicząca! szanowni nie możemy na ευχαριστώ και Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση των βασικών κανόνων του πολιτισμού στην Καμπότζη. Υπάρχει τεράστια πολιτική καταπίεση. Κόσμος συλλαμβάνεται επικεφαλής της αντιπολίτευσης πρόκειται απλά για βαρβαρότητα δεν είναι πολιτική διαμάχη αυτή ε, καταστρέφεται η αντιπολίτευση με τρόπο βάρβαρο πρέπει να αντιδράσουμε με τον τρόπο που κάνουμε πριν από 20 χρόνια στις πρακτικές των κομμουνιστικών καθεστώτων όταν συνέβαιναν τα ίδια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το ψήφισμα. Και κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Πάρα πολλά εξαρτώνται από την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να εξαρτηθεί από την τήρηση αυτών των προδιαγραφών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Κοράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, οι κατάφορε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταστολή που βλέπουμε ανελαμβάνει χώρα στην Καμπότζη θα μπορούσαν να συνεχιστούν με τη συγκατάβαση που μέχρι τώρα έχει επιδειχθεί ω προς την ε, πολιτική της Καμπότζης. Όμως και από του επενδυτέ υπάρχει τι πολυεθνικές, υπάρχει μεγάλη τάση κερδοσκοπία. Στην Καμπότζη η χώρα βρίσκεται σε πώληση. Τα δάση, οι λίμνε το πετρέλαιο, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των 700.000 ανθρώπων που εκτοπίστηκαν για να γίνουν επενδύσεις στην γεωργία, για την αρπαγή γεών, τα δικαιώματα των εργατών, των παιδιών, των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της ένδυσης και ουσιαστικά στέλνουν τα προϊόντα στη δική μας αγορά. Εδώ δεν έχουμε ποτέ ε, λάβει μια θέση ισχυρή και με πυγμή. Το ψήφισμα αυτό ε, δείχνει ότι έφτασε η στιγμή να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέντα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα από πλευρά ε, του ΕΛΚ να εκφράσω τι ανησυχίε μα σε σχέση με την κατάσταση στην Καμπότζη λόγω τη βία ε, κατά βουλευτών, ένταλμα σύλληψη για τον ηγέτη τη αξιωματική αντιπολίτευση ε, Είμαστε σε ένα σημείο καμπή στην Καμπότζη. Μην ξεχνάμε ότι είναι και μεγαλύτερο εταίρο μας ως προς ε, την αναπτυξιακή βοήθεια. 410 εκατομμύρια έχουν προβλεφθεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Απευθύνουμε και δοκιμάτων σε έναν απελευθερώσει κρατουμένου που κρατούνται παράνομα να αποκαταστήσει τα, την ασυλία τους ουλευτική ασυλία τους και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα της ε, κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, ο επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υποπέδει την κατάσταση στη χώρα. Σας ευχαριστούμε η Σεσίλια Βίκστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μου είναι ιδιαίτερα αγαπητή η Καμπότζη και πραγματικά είναι ιδιαίτερα επώδυνο όταν βλέπω πόσο αυξάνεται η επιθετικότητα και η βία της κυβέρνηση κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 11 κρατούμενοι και πολιτικοί κρατούμενοι δεν έχουν δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Είναι μεγάλες ε, οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί και δεν υπάρχει καμία θεμητή αντιπολίτευση. Ο Σαμ Ρένσι ε, έχει, ε, κρατείται κατοίκο και κατηγορείται για παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. το αντίθετο συμβαίνει διότι είναι θεμητός ηγέτης της εξωματικής αντιπολίτευσης. Παρόλα αυτά δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης. Το, δίκαιο, το κράτος δικαίου έχει πολιτικοποιηθεί και τα μέλη της αντιπολίτευσης διώκονται. Χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίνουμε το σημερινό ψήφισμα, διότι η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της έκθεσης είναι ένα καθολικό δικαίωμα, ενώ συστηματικά η κυβέρνηση της Καμπότης καταπατά αυτά τα βασικά δικαιώματα. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν για το ψήφισμα, διότι είναι σημαντικό για τη δική μας την αξιοπιστία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ. Η πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη υποβαθμίζεται διαρκώς, ιδίως από τις 13 Νοεμβρίου, όταν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στις 13 ε, Νοεμβρίου και ήρθε η βουλευτική του ασυλία. Επίσης, ακτιβιστές της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν ποινές κάθεξης μεταξύ 7 και 10 ετών. Επίσης μια ομάδα διαδηλωτών κατά τη κυβέρνησης δέχτηκε άγρια επίθεση και δύο βουλευτές ε, συγκεκριμένα από την αντιπολίτευση ήταν μέλη αυτής της ομάδας. Πρέπει λοιπόν να υψώσουμε τη φωνή μας και πρέπει όλοι οι ακτιβιστέ και τα μέλη της Εθνικής τη Γερουσίας που δέχονται πολιτικές πιέσεις να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ελεύθερα. Εδώ η κυβέρνηση θα πρέπει να πάβει να διώκει του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξασφαλίσει κατάλληλε συνθήκε η απελευθέρωση όλων των πολιτικών ε, κρατουμένων με επινοημένες κατηγορίες ως επιτοπλίστων. Ευχαριστούμε για η κυρία Βεζιά. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά συμμετείχα σε συνεδρίαση της αντιπροσωπείας για το συντονισμό των εκλογικών ε, των ε, αποστολών εκλογικών παρατηρήσεων. Η Καμπότζη μα ανησυχεί στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Τον Ιούλιο καταγγείλαμε τον νόμο για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και την ε, κατάσταση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα ανεργίας των νέων πάνω από 50% και ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν ε, πέσει θύματα της αρπαγής γεών προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών ε, που παράγουν τρόφιμα και τα πράγματα αυτά διαρκώ επιδεινώνονται. Η πολιτική κρίση ε, επιδεινώνεται διαρκώ μετά τι εκλογέ του Ιουλίου του 2013. Διώξει ασκούνται καθημερινά στου αντιπολιτευόμενου και σε όλου του στρατευμένου κατά τη κυβέρνηση το ίδιο και για τις ενώσεις και συλλόγους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Καμπότζη να δεσμευτεί στον δρόμο του διαλόγου πριν υποβαθμιστεί και άλλο αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να δεσμευτεί με τις διεθνείς της υποχρεώσεις η χώρα αυτή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λοκ Μπίλερ δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Οπότε προχωρούμε. εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Ζητούμε την κατάσταση στην Καβότζη και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι έχει εγκριθεί νομοθεσία κατά του ιδιωτικού τομέα, κατά της κοινωνίας των πολιτών που δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ και διαφόρων ενώσεων οργανισμών και σωματείων. Δυστυχώς η κυβέρνηση και η Βουλή της χώρας αγνόησε τα σχόλιά μας και ε, πέρασε αυτή την νομοθεσία. Δυστυχώς η Καμπότζη παρόλο που είμαστε ο βασικότερος εταίρος της αγνοεί τα όσα λέμε στα ψηφίσματά μας και εκατοντάδες ε, εκατομμύρια ε, δίνουμε στην ανάπτυξη της χώρας αυτής και στο προσεχές μέλλον. Θα δώσουμε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανασκεφτεί αυτή την προθυμία μας ε, να βοηθούμε εφόσον μας αγνοεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιτεν Χαλτσαρ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η Καμπότζη είναι από τις πιο δοκιμαζόμενες χώρες και δοκιμασμένες στην Ένωση. Τα εγκλήματα ε, του καθεστώτος Πολ με εκατομμύρια θύματα ακόμα ρίχνουν τη σκιά τους στη χώρα. Είναι δύσκολο να επανέλθει στην νομιμότητα. Έχει παλινοδίες ε, και ε, πέρυσι είχαμε περιορισμό της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και τώρα αυτό έχει φτάσει μέχρι τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Αυτό έχει να κάνει και με τον ηγέτη ε, της αντιπολίτευσης της Δημοκρατικής που είναι δημοφιλής και αυτό ε, δημιουργεί εκνευρισμό στην κυβέρνηση είναι στην εξορία και παρευρίσκεται για τις αντιπολίτευσης εδώ σήμερα στο θεωρείο και προς όφελος όλων θα ήταν να βρίσκεται σήμερα στην Πνόμ και στη Βουλή της Καμπόζης, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το επιθυμούμε όλοι και γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποστηρίξει και καλούμε και την κυβέρνηση της Καμπότζης για να βγει από το σκότος της ιστορίας οριστικά αυτή η χώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Χαιρετίζουμε και εμείς τον κύριο Άντσι και δίνω το λόγο στον κύριο Γιάκοφτσιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 στο 2020 θα βοηθήσει με αναπτυξιακή βοήθεια την Καμπότζη της τάξης των 410 εκατομμυρίων ευρώ. σε ένα καθεστώς καταπιεστικό ε, που καταστέλει τις ελευθερίες ε, ε, και φυλακίζει τους αντιπάλους. Είναι από τις πιο φτωχές χώρες. Η οικονομική πολιτική κατάσταση βυθίζεται στην καταστολή. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αντιδράσουμε και εγώ υποστηρίζω για το λόγο αυτό το ψήφισμά μας. Είναι ένα σαφές μήνυμα που στέλνουμε στις αρχές της χώρας αλλά και στην κοινωνία των πολιτών ότι είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε και λέμε ξεκάθαρα ότι δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση που είναι απαράδεκτη και ζητούμε αλλαγέ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και τη δημοκρατική αντιπολίτευση. Η πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματο του αυτού του συμμεμονωμένοι <laughs> ομιλητέ, ο κύριο Σάμπα Σόγκορ. Ευχαριστώ. Ε, ο πολιτικός βίος της Καμπότζης αυτή τη στιγμή πρέπει να οδεύσει σε ένα σημείο που τα δύο, τα δύο κυβερνώντα στρατόπεδα θα έρθουν σε διάλογο μεταξύ τους. Ε, θα πρέπει να δούμε τη στάση της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή καταστέλει την αντιπολίτευση και τον δημοκρατικό ανταγωνισμό και σε αυτό το σκηνικό θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις πιστεύω, ιδίω επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποδώσει 410 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή βοήθεια προς την Καμπότζη. Είμαστε ο πρώτος μεγαλύτερος εταίρος της Καμπότζης. Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον θέλουμε να προστατεύουμε τις αξίες μας σε όλο τον κόσμο, να είμαστε σαφείς στην αναπτυξιακή μας πολιτική, να θέσουμε και τέτοια κριτήρια. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θέλω να επικεντρωθώ στην πολιτική κατάσταση, συμμεριζόμενος όσο είπαν και οι συνάδελφοι, κυρίως για την αρπαγή των γεών. Η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή προβλέπει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά χωρίς δασμού, αλλά αυτό είχε δραματικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό, ιδίως λόγω του φαινομένου ότι βία ε, διώκονται οι αγρότες από τις περιοχέ τους για να περιέλθουν στα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων ε, οι εκτάσει αυτές όπως η Delta Line της Μεγάλης που εν μέρει είναι υπεύθυνη και δεκάδες χιλιάδε ε, στρέμματα γης αρπάζονται από τους χωρικούς. Εδώ λοιπόν η Επιτροπή είχε απαντήσει σε ερώτησή μου ότι θα πρέπει μια διαμέσα αναθεώρηση τον Νοέμβριο του 2017 και μπλα μπλα, αλλά όλα αυτά είναι φλιαρίε. Ε, κυρία Επίτροπε, είσαστε μέλο του Κολεγίου των Επιτρόπων. Θα πρέπει να δούμε εάν όντω τα δικαιώματα μπαίνουν πριν από την, ε, το εμπόριο. Και εάν θα παρακολουθούμε σωστά ή ενδεχομένω θα διορθώσουμε τι συμφωνίε που έχουμε ήδη συνάψει. Ευχαριστούμε φαίνεται ότι είμαστε εντός των χρονικών ορίων, οπότε θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους με τη διαδικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ευχαριστώ. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, πιστεύω και εγώ πως θα έπρεπε να επενεξεδώσουμε την κατάσταση στην Καμπότζη. Λαμβάνοντα υπόψη ότι είναι πολύ υψηλό το ποσοστό της αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουμε σε αυτή τη χώρα, οφείλουμε να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Δέχονται αυτή την αναπτυξιακή βοήθεια και άρα θα πρέπει να δέχονται και την πίεση που ασκούμε στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ελευθερία για τους πολίτες, να λειτουργεί ελεύθερα η αντιπολίτευση, να, ε, να γίνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών. Αλλιώς θα πρέπει να επανεξετάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνουμε στην Καμπούτση για να ασκήσουμε ακόμη περισσότερη πίεση στην κυβέρνηση για να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές. Ευχαριστώ, ο κύριος Ντονάνο. Ευχαριστώ. Όντω, ε, διαφθορά και πελατειακό κράτο είναι χαρακτηριστικά πολιταρχικών ε, καθεστώτων. Είναι καθήκον μα ε, παντού όπου χρειάζεται να αγωνιζόμαστε κατά αυτών των πρακτικών, κυρίω όταν του δίνουμε και αναπτυξιακή βοήθεια. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτική κρατούμενη είναι απαράδεκτε πρακτικέ για εμά του Ευρωπαίου. Με μια φωνή θα πρέπει να υπερασπιστούμε την δημοκρατία στην καμπότσια, όπως και σε όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου είναι βασανισμένη η χώρα, ταλανισμένη από την ιστορία. Πρέπει να τη βοηθήσουμε να ξαναβρει το δρόμο της δημοκρατίας. Επίτροπε, θα πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος με την κυβέρνηση για να εξακριβώσουμε ακριβώς πώς χρησιμοποιείται η αναπτυξιακή μας βοήθεια, ότι χρησιμοποιείται όντως για την ε, αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην Καμπότζη το καθεστώς του Χουν Σεν που βρίσκεται στην εξουσία για πάνω από τριάντα χρόνια έχει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ημερήσια διάταξη. το ίδιο ισχύει και για την έλλειψη πολυφωνίας και τη φήμωση και τις διώξεις κατά της αντιπολίτευσης. ταυτόχρονα οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας δρούν ανεξέλεκτα καταστέλλοντας διαδηλώσεις και απεργίες. στο οικονομικό πεδίο η χώρα μαστίζεται από τη φτώχεια παρότι η καμπότζη είναι πλούσια χώρα με ορυχεία ξυλία πετρέλαιο και όμως ο λαός της καμπότζης δεν έχει καρποθεί τα έσοδα από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με κύριο στοιχείο τη διαφθορά και τη διαπλοκή των πολιτικών και των επιχειρηματιών. το 45 του εδάφους της χώρας έχει παραχωρηθεί για τους δίθεν επενδυτές ενώ από το 2003 περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από τη γη τους και το 14% της συνολικής γης έχει χαθεί από τα χέρια των μικροκαλλιεργητών εν ώψη της αναπτυξιακής βοήθειας που δίνει η ευρωπαϊκή ένωση στην καμπότζη πρέπει να ασκηθεί πίεση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ ε, για την παρουσία του ηγέτη της αντιπολίτευσης Καμπότζης, που είναι και μέλος της... Ε, ε, συνοδεύεται μάλλον από μια βουλευτή. Σας καλωσόριζω και τους δύο. Είναι σαφές το ότι το Χουντσέν θα πρέπει να σταματήσει την καταστολή και την δίωξη της αντιπολίτευσης και να σέβεται το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο μας καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές. Καλούμε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει τις business as usual με την Καμπότζη. Είμαστε ο πρώτος δωρητής. Καλούμε τον Χουνγκ Σεν και ε, την κυβέρνησή του να αφήσει ελεύθερο τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και να αποκαταστήσει την κοινοβουλευτική του ασυλία. Η δημοκρατία και η μη βία τελικά θα επικρατήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τρεμόσα. Ο κύριος Πόλτσακ, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η δική μου άποψη είναι ότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η αναπτυξιακή βοήθεια που προσφέρουμε προς την Καμπότζη συνδέεται με το κατά πόσον σέβονται τις δικές μας απαιτήσει. Έχουμε γκρίνει και στο παρελθόν ψηφίσματα, ίσως ούτε καν μόνο ένα, που καλεί καλούν την Καμπότζη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Είναι μια χώρα ομοιογενής ως προς τον πληθυσμό της και την θρησκεία της. Πρόκειται για μια κοινωνία με συνοχή, κατά την άποψή μου λοιπόν. Δεν πρέπει αυτή η ομογένεια να μετατοπιστεί σε άλλους τομείς όπως αυτός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε και τον οικοκυριό μα πρωτού καταδικάζουμε του άλλου. Οι εταιρείε που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που φελούνται τη κατάσταση στην Καμπότζη, ε, εκμεταλλευόμενοι την απελπισία των κατοίκων, είναι ένα βασικό πρόβλημα. Σα ευχαριστώ. Φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ε, Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας, όντως. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γεωργίευα. Έχετε το λόγο κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ. Από της Αντιπροέδρου και υψηλής είπα τη εκπροσώπου, ο κ. Μογκερίνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους βουλευτές ε, που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Οι πρόσφατες κινήσεις κατά των μελών της αντιπολίτευσης στη Καμπότζη που περιέγραψαν προλαλήσαντες ε, με κάθε λεπτομέρεια, όντως συνιστούν πηγή σοβαρών ανησυχιών και γύρουν ζητήματα σε σχέση με το διάλογο ε, που συμφώνησαν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πέρσι τον Ιούλιο. Δεν χρειάζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος ε, μια, της αντιπολίτευσης ε, στα δημοκρατικά δρόμενα. Είναι η φύση, εκφύσεως έχει την ευθύνη η, αντιπολίτευση να ε, φροντίζει το ώστε να λογοδοτεί η κυβέρνηση. Η Καμπότζη έχει υποστηρίξει αυτό τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα στα δύο βασικά κόμματα της ε, Καμπούτζη και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται η αντιπολίτευση από το να διαδραματίζει αυτόν τον θεσμικό της ρόλο. Δεν θα πρέπει να καταστρέφεται, να μπορεί να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να μην ε, να απαγορεύονται οι προσωπικές επιθέσεις κατά μελών της αντιπολίτευσης. Είναι σε θέση ισχύω ε, η κυβέρνηση και γι' αυτό έχει καθήκον να αυτό περιορίζεται να δρά υπεύθυνα. Να, δρά να υπάρχει εμπιστοσύνη και ε, με υπομονή να συνεχίζεται ο πολιτικός διάλογος. Είναι σημαντικό για την Καμπότζη, για την ίδια τη χώρα να επιστρέψει στην οδό της συνεργασίας, της δέσμευσης ως προς τη δημοκρατική κοινωνία. Επανειλημμένα έχουμε εκφράσει ανησυχίες μας σε σχέση με τις επιθέσεις ε, κατά δύο βουλευτών και δια της διπλωματικής οδού ε, Απευθύνουμε διαρκώς εκκλήσεις στα δύο βασικά κόμματα να επιστρέψουν σε, αυτή την, σε αυτό το πολιτικό διάλογο που είχαν συμφωνήσει πέρσι τον Ιούλιο. Ποιε είναι οι εναλλακτικέ για την πολιτική. Αυτό πρέπει να είναι το αντικείμενο του πολιτικού διαλόγου. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί και να συνεχίσει να προοδεύει αυτή η χώρα. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, και την αναπτυξιακή μας βοήθεια συγκεκριμένα τα 410 εκατομμύρια για την καλή διακυβέρνηση ε, στην Καμπότζη για να υποστηρίξουμε και εμείς αυτή την διαδικασία εκδημοκρατισμού. Σας ευχαριστούμε κυρία Γεωργίευα. Θα θέλαμε